Εγκρίνεται. Τροπολογία 50-55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 50-57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η ίδια πλειοψηφία. Τροπολογία 50-66 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 50, 92 υπέρ. Α, συγγνώμη, λέει πρόεδρος, ήταν η 50-67 πρώτα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα τροπολογία 50-92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50-93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50-94 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Μήπως μπορούμε από την 50-95 μέχρι και την 50-97 μαζί. Αυτές τις τρεις τροπολογίες μαζί λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 50 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 50-99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51-00 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50-31 υπέρ, κατά, αποχές, θα επαληθεύσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 51-01 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50-77 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 51-24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 51-03 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51-04 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51.05 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συγγνώμη, λέει η πρόεδρος, απορρίπτεται. 50.30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50.28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5106 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5005 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5125 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5062 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51-21. Εδώ έχουμε προφορική τροποποίηση. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50-65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50-21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5012, 12 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Αποχές, διορθώνει ο πρόεδρος, εγκρίνεται. 51-07 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50-25 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 δεκατρία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50-33. 5033 33 υπέρ. Κατά. Α, μια στιγμή, μια στιγμή. Λέει πρόεδρος, πρώτο τμήμα, γιατί είναι κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα της 5033 33 υπέρ. Κατά. Το πρώτο τμήμα απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50-34 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. 50-34. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 50-68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51-29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51-28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50-75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5079 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5087 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5108 υπέρ, κατά, αποχές, α, θα ελέγξουμε εδώ ηλεκτρονικά παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 50, 80 και 50, 58 γιατί είναι ίδιες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 50, 01. Καταπίπτει. 50-74. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50-59. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50-73 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50-81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50-06 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50-60 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 50-72 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 50-04 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5071 Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 5016 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50-70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50-08 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51-30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50-84 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50-09 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51-31 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 51-32 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα έχουμε τη συμβαστική τροπολογία αριθμός 1 και θα δώσω το λόγο στην κυρία Μουνίθ η οποία θα κάνει μια διόρθωση. Ευχαριστώ. Έχουμε μια συμβαστική τροπολογία που επισυνάπτεται στον κατάλογο ψηφοφοριών. Είναι μια τροπολογία ε, επί των παρατηρήσεων και έχει ως εξής. Ένα τμήμα των υποχρώσεων αυτών, τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει αποκλειστικά να αφιερωθεί στη χρηματοδότηση ε, της εκκίνησης του σχεδίου του πενταετούς για phasing out, για να καταληφθούν δηλαδή οι καλλιέργειες όπιων προκειμένου να έχουμε ε, μια πραγματική αλλαγή σε αυτό το τομέα, σύμφωνα με τη, όσα έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή του μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν που εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 2010. Κυρία Μουνίθ. Το ποσό νομίζω ότι πρέπει να το αλλάξετε, γιατί στον κατάλογο ψηφοφορίας το ποσό που δίνεται είναι σφαλμένο. Α, ναι, ναι, λέει κυρία Μονίθ, πρέπει να διορθώσω. Είναι λάθος τα ποσά που αναφέρονται στον κατάλογο ψηφοφορίας. Στην πρώτη στήλη, στις υποχρεώσεις, πρέπει να βγάλουμε το 3. Είναι 5.085.000. 5.085.000 και στις πληρωμές είναι 18 εκατομμύρια. Μεγάλη διαφορά, λέει πρόεδρος. Καλώς. Κύριε Σαλαφράγκα. Α, συμφωνεί το ΕΛΚ. Ωραία, καλώς. Οπότε, συμβιβαστική τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51-22. Όχι, περνάμε στην 51-26. Σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 51-27 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στην 5085 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τα χέρια είναι όλο και πιο αραιά. υπέρ κατά αποχές δεκτή. 50-63 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 50-13 και 50 που ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 50-61 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 50-64 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, <clears throat> κατά, αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50, 14 και 50, 78 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 5069 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 50-38 υπέρ να κάνουμε μια ομαδοποίηση τροπολογιών. Οι τροπολογίες αυτές έχουν μια προφορική τροπολογία εδώ για ένα ποσοστό αποθεματικό, λέει ο κ. Γουαλτιέρη. Λοιπόν, θα πάρουμε από κοινού από την 5038 όλες οι τροπολογίες Γκουαλτιέρη μέχρι την 5049. Συμφωνείτε? Ποιος είναι υπέρ των τροπολογιών Γκουαλτιέρη? Κατά αποχές εγκρίνονται. 50-20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50-36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50-24 ε, εκπίπτει, 50, 50 γκολτιέρι. Μπορούμε και εδώ να κάνουμε μια ομοδοποίηση. Μέχρι την 50-54 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτες δεκτές. 5-29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συγγνώμη, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 529, Παρακαλώ, άρχεται. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Δεν υπάρχει τελική ψηφοφορία, λέει η πρόεδρος. Τελείωσε η διαδικασία λοιπόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την κυρία Μινίθ. Η επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας, 17 Σεπτεμβρίου, για ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του Κουσιφού Πεδίου. Οι συντονιστές μπορούν να παραμείνουν στην αίθουσα, θα έχουμε μία μικρή συνεδρίαση του